Colleagues, Κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ε, σας, αναφέρω ότι έγινε... Έχετε πάρει τα πρακτικά της συνεδρίας των συντονιστών εχθές, ως συνήθως, οπότε περνάμε στο σημείο 12. Έχουμε ψηφοφορίε. Και ξεκινάμε με την ε, έκθεση του Γιάννη Ζαντό για τη διεθνή εμπορική πολιτική στο πλαίσιο των επιταγών της αλλαγής του κλίματος. Θα πάμε μία-μία της τροπολογίες. Έχετε όλες τις κάρτες σας. Okay. Everything's okay? So let's start the vote. Amendment... Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. You Τέλο vote ψηφοφορίας. Απορρίπτεται όντως. Το αρχικό κείμενο, παράγραφος 1, χωριστή ψηφοφορία έχει ζητηθεί. Πρώτο τμήμα. της παραγράφου 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. amendment 16. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Amendment 17, there's an oral amendment. Τροπολογία 17. Υπέρ. Ε, υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά? Όχι. Ε, ποιος είναι ο συντάκτης της προφορικής τροπολογίας? Ο κύριος Γκλάτφελντερ. And uh, it consists of uh, replace Replace the word supporting by subsidizing. Αντί για supporting να λέει subsidizing. Those in favor. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18.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 Σοσιαλιστές και πράσινοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε, δεν είμαι βέβαιος. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ανθρωπολογία 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Χωριστή ψηφοφορία. Υπέρ. Του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. υπέρ, κατά, αποχές, εγκλίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ, Κατά. Αποχές. Δεν είμαι δεν σας ελέγξουμε. Vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την παράγραφο 3. Τέλος της ψηφοφορίας. Adopted. Um, amendment 21. Τροπολογία 21. Χωριστή ψηφοφορία. Προφορική τροπολογία που βρίσκεται. 21. Η αντικατάσταση της λέξης ΠΟΕ από το διεθνείς κανόνες. Διεθνείς κανόνες αντικαθιστά το ΠΟΕ. Αυτή είναι η τροπολογία, η προφορική. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας ψηφίσουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 20, ή μάλλον τροπολογία 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 24 έχει καταπέσει. Ωραία. 25. 25 τώρα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Paragraph 9. Paragraph 9, original text. Παράγραφος 9. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Τροπολογία 32. Αντιρρήσεις για προφορική τροπολογία, όχι. Παρακαλώ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Η προφορική τροπολογία είναι να διαγραφεί η λέξη perverse. Καλή την Κομισιόν ε, ώστε να επαληθεύσει ότι δεν θα δημιουργηθούν ε, μη επιθυμητές επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές απορρίπτεται. Τριάντα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Ας το επαναλάβουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό παρακαλώ. Check. Έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 34. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πρωτότυπο κείμενο της παραγράφου 19 χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 39, υπέρ. Αποχές, εγκρίνεται. 40, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41, υπέρ. Against κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αρχικό κείμενο παράγραφος 43 Παράγραφος 23, με συγχωρείτε, χωρίς την ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, παράγραφος 24, τροπολογία 43, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 44, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 25, η ομάδα ECR έχει ζητήσει χωριστή ψηφοφορία σε πέντε τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.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 Παράγραφος, μάλλον τροπολογία 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 29, χωριστή ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ναι, να το ελέγξουμε, ναι. 48. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός έλεγχος. The vote is closed. Rejected. Amendment 49 in favor. Τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 31. Χωριστή ψηφοφορία. Τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο της παραγράφου 22. Ε, και πάλι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 απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, τα εκτιμώντας 1, α, συγγνώμη, τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστικές τροπολογίες 1. Ε, στο εκτιμώντας β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αρχικό κείμενο του δεύτερου εκτιμώντας, χωριστή ψηφοφορία. False. False. False. False. false. Α, όχι, έχει καταπέσει. Τροπολογία 4. You are right. Amendment number 7. Τροπολογία 7. Χωριστή ψηφοφορία. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Γιατί εκτιμώντα γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπάρχει προφορική τροπολογία στην 12 υπάρχουν αντιρρήσεις για προφορική τροπολογία η προφορική τροπολογία λοιπόν θα αντικαταστήσει το τελευταίο τμήμα της τροπολογίας θα αντικαταστήσει το end από το but και θα λέει ότι ο χρόνος προσωπεύεται καλύτερα και θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο του εκτιμώντας ε χωριστή ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Δεν είμαι βέβαιος για το αποτέλεσμα. Δεύτερο τμήμα του πρωτότυπου κειμένου στο εκτιμώντας ε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος πληροφορίας Εντάξει, εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τέλος. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογίες της Επιτροπής Ανάπτυξης. No, if you wish, if they Any, any objections? Any objections to a block vote of Deve's amendments? Θέλετε να ψηφίσουμε μπλόγκο όλε τι τροπολογίε. Όχι, υπάρχουν αντιρρήσει. Οπότε α ψηφίσουμε χώρια. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται.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 αισθάνομαι κάπω σαν τον κύριο Σούλτσα στην Ολομέλεια. Αλλά θέλω να ενημερώσω την ομάδα μου ότι καλό είναι να απέχουμε. Ναι, ο Σούλτσα τα λέει αυτά συνήθω στην Ολομέλεια, έτσι δεν είναι. Ωραία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεση όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίνεται 14 υπέρ, 4 κατά και 8 αποχές. Now let's move to the of the Ας περάσουμε λοιπόν στο σχέδιο έκθεσης της ε, Τόκια Σαΐφη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά και περιβαλλοντολικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Περνάμε λοιπόν στην τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμόν 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παίρναμε λοιπόν στην επόμενη, η οποία είναι η 36η. Τροπολογία 36 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική υπαριθμό 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 53, περνάμε στην 53, υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. Uh, Περνάμε λοιπόν στην 53. Ωραία. Έλξη ψηφοφορία. Ωραία. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την 56. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 64. Πάμε στην 64. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν. Let's move to the of the recite. Να ψηφίσουμε λοιπόν τώρα και τα εκτιμώντας. Περνάμε στο νέο εκτιμώντας ΑΑ. Είναι μια προφορική τροπολογία. Α, ξέχασα, με συγχωρείτε, καταρχήν την τροπολογία 7 που είναι το εκτιμώντας α. Το 7 λοιπόν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα σε ένα νέο εκτιμώντας που είναι το ΑΑ, είναι προφορική τροπολογία, έχουμε αντιρρήσεις. Ωραία, ας ψηφίσουμε λοιπόν, η προφορική αυτή ε, τροπολογία βρίσκεται ε, στα φάκελο μπροστά σας, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία νούμερο 10. Α, για την ενάτη. Θέλουμε να κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Για την τροπολογία 9 θα κάνουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Απορρίπτεται. Σας παρακαλώ πολύ να σηκώνετε τα χέρια σας. Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη. Είναι η υπαριθμό 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές Μάλιστα, δεν εγκρίθηκε η τροπολογία υπαριθμών 10, άρα θα πρέπει να ψηφίσουμε και την υπαριθμών 11. Κάνετε, έχετε δίκιο που μου το υποδεικνύετε. Περνάμε λοιπόν στην 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα πάμε στη συμβιβαστική υπαριθμών 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 12η έχει αποσυρθεί. Περνάμε λοιπόν στο εκτιμώντα δέλτα, όπου έχουμε μια προφορική τροπολογία. Έχουμε εδώ αντιρρήσει στην προφορική αυτή τροπολογία. Α την ψηφίσουμε υπέρ προφορική υπαριθμών 2. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην επόμενη που είναι η 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Σε 15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στη 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Στη 17 εδώ έχουμε χωριστεί ψηφοφορία στο πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται και στο δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές. Για να το δούμε ηλεκτρονικά για το δεύτερο τμήμα της 17, παρακαλώ ξεκινάει η ψηφοφορία και λίγη. Απορρίπτεται. Η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβιβαστική υπαριθμών 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Uh, amendment number 3 in Για την 3 υπέρ. Κατά αποχές ή 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή έξι υπέρ α, κατά και αποχές και εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στις τροπολογίες που έχει υποβάλει η Επιτροπή ΑΦΕΤ εξωτερικών υποθέσεων. Περνάμε τώρα στην παράγραφο 6, υπέρ, κατά, αποχές, γκρίνεται. Στην 8, υπέρ, παράγραφο 8, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 14 σε χωριστή ψηφοφορία σε δύο τμήματα, στο πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πηγαίνουμε στη 15 υπέρ, κατά, αποχές. Για να δούμε ηλεκτρονικά. Για τη 15 θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινά η ψηφοφορία. Έλεξη ψηφοφορία απορρίπτεται. Amendment 17 in favor. Υπέρ στη 17. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. let's vote 20, yes. Ή 20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. επόμενη είναι αυτές που έχει υποβάλει η Επιτροπή Απασχόλησης, η 6 και η 7, με συγχωρείτε, η 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 7 τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στη 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Στην 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει με τον αριθμό των ομάδων, γιατί νομίζω ότι στο ΕΛΚΑ έχουμε 11 και όχι 10. It would appear here if there is any extra vote, so we don't have any record on that. Apparently everything... Δεν έχουμε βρει κάποια ψήφο παραπάνω, οπότε ευχαριστώ που μας το υποδεικνύετε, αλλά δεν έχουμε διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Of envy. Uh, amendments... Πάμε λοιπόν στις τροπολογίες από την Επιτροπή ΕΝΒΗ, στην 6 Στην 6 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στη 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περιμένουμε στις τροπολογίες που μας έχει υποβάλει η Επιτροπή ΔΕΔΕ. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 2. 2 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να επαναλάβουμε σας παρακαλώ πολύ διανατάσιο στις χειρός είμαστε στην ΔΕΗ 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 4 υπέρ κατά Άποχες. Απορρίπτεται. Παράγραφος 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στην 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7. Η 7 καταπίπτει λοιπόν. Περνάμε στην 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Στη 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Για την έκθεση αυτή με τις τροπολογίες που εγκρίναμε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίθηκε με 22 υπέρ, 2 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια για την επιτυχημένη αυτή προσπάθεια. Let's move to the vote of the... Για να περάσουμε λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω από τον Πρόεδρο να επιταχύνει λίγο την ψηφοφορία, γιατί έχουμε ψηφίσει δύο εκθέσεις μέσα σε μία ώρα. Ε, δεν είναι και κάποια εξαιρετική επίδοση για την Επιτροπή μας αυτή. Νομίζω μπορούμε να πάμε και λίγο πιο γρήγορα. Εγώ θα προσπαθήσω, αλλά εσείς σας παρακαλώ πολύ, όταν ζητάω να ψηφίζετε, να σηκώνετε το χέρι σας. Και την επόμενη φορά ε, οι λιγότερες τροπολογίες. Αυτή είναι η άλλη λύση. Γιατί κοιτάξτε τι έχω εδώ πέντε τροπολογίες έχω εδώ για αυτή την έκθεση. Τι νομίζετε δηλαδή, εσύ ότι μπορούμε να τα κάνουμε σε 5 λεπτά. Εγώ σας προσφέρω τη θέση μου. Θέλετε να κάνουμε τι είδου ψηφοφορίε για να τα κάνουμε γρήγορα. Να περάσουμε λοιπόν για την κοινωνική εταιρική ευθύνη την επόμενη δηλαδή, για να δούμε και τον τίτλο. Amendment number one, in favor. Πρώτη, υπέρ, κατά. Δύο, εγκρίνεται. Πέντε, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Η 47, υπέρ, κατά αποχές καταπίπ... Ε, ε, απορρίπτεται. Στην 47 ξεκινάει η ψηφοφορία. Λίγη. Ωραία. Στην 48 λοιπόν χωριστή. Υπέρ για το πρώτο τμήμα. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται για το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές για να το δούμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 52 ωραία ξεκινάει η ψηφοφορία λίγη απορρίπτεται συμβιβαστική υπάρχουν 5 υπέρ Συμβιβαστική 5, σας παρακαλώ πολύ. Όχι 5, με συγχωρείτε. Yes. 53. Ε, στην 53 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 57 υπέρ, κατά, αποχές. Και δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το αποτέλεσμα. Στην 57 παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. The vote is closed. Λίγη. And result is... Και απορρίπτεται. Ακολουθεί η τροπολογία 58, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. 63. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Ισοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. τρία υπέρ. Εβδομήντα τρία. Υπέρ λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75 υπέρ. Α, α, ζητείτε επαλήθευση για την 74. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει. Απορρίπτεται με ψηφία. 75 λοιπόν τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Υπαριθμόν 9. Α, ζητάτε επαλήθευση της ψηφοφορίας για την 76. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται και αυτή Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84. Αυτή εκπίπτει. Συμβαστική υπάρχουν 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Α. Ζητείτε επαλήθευση για την 90. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ζητάτε λοιπόν επαλήθευση της 91. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές δεν μπορώ να είμαι βέβαιος ας επαληθεύσουμε 94 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και αυτή. Ακολουθεί η παριθμόν 96 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται 98 υπέρ. Καλώς σα επαληθεύσουμε την 97, αφού μου το ζητείτε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Α, πρώτα η 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 100. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 101. Υπέρ. Κατά. Κατά. Κατά παρακαλώ. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση 101. Αρχίζει. Πέρας. Α, εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 102 υπέρ. Κατά. Ψηφίσατε όλοι. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. 102. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε επαλήθευση για την 103. Καλώς. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται αυτή. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Νέα αιτιολογική σκέψη παριθμών 11 τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δώδεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά <clears throat> αποχές εγκρίνεται. Όχι λέει ο πρόεδρος. 17. Ας επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. Συμβιβαστική. Συμβιβαστική τροπολογία υπάρχουν 2. Υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ, σηκώστε καλά τα χέρια. Συμβαστική 2 λοιπόν, υπέρ, κατά, εποχές,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 25 υπόρ, υπέρ, συγγνώμη, κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή. 27 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αν καλώς, επαλήθευση για την 28, αρχίζει. Λείπει μία ψήφος. Πέρας. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κάτα. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική παριθμών 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 προφορική του ίδιου του εισηγητή. Έχει κανείς ένσταση. Όχι, ψηφίζεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Συμβαστική υπαριθμών 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παραθέσεις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 δηλαδή η δέλτα, J και η παράγραφος 10. Συμφωνείτε με την πρόταση αυτή να ψηφιστούν όλες μαζί. Πώς να προχωρήσουμε πιο γρήγορα τότε. Όλες λοιπόν μαζί τις αιτιολογικές σκέψεις. Όλες, εκτός από τις δύο που καλύπτονται ήδη. Όλες λοιπόν τις υπόλοιπες μαζί, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Η παράγραφη τώρα. Ένα. Δύο. Συγγνώμη. Αποχές. Κατά. Εγκρίνεται. Δύο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τέσσερα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 Πέρας. Εγκρίνεται λοιπόν. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Α, καλύπτεται η ναι, Σωστά, σωστά. Η 11 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτή. Τελική ψηφοφορία θα γίνει ονομαστική, δηλαδή με ηλεκτρονικά μηχανήματα. Αρχίζει. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Συγχαρητήρια. Αγαπητέ Αρλέμ Ντεζίρ. Moving <coughs> item 15 is... Το 15 θέμα έχει αναβληθεί. Τελειώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Μα ήταν πραγματικά εκατοντάδες οι τροπολογίες. Ας προχωρήσουμε τώρα στο 18, 19 και 20 που θα τα συζητήσουμε όλα μαζί. Παρακαλώ. Όσοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα, να το πράξουν ησυχώ. Keeping... Όσοι εξακολουθούν να συζητούν, στα νεοελληνιστή αποκαλούμενα πηγαδάκια, παρακαλούνται και αυτοί να εξέλθουν. Παρακαλώ, σταματήστε τις συζητήσεις. So, points 18, 19 and 11. 18, 19 και 20 λοιπόν μαζί συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Βασιλείου του Μαρόκου για την, επίλυση για την θέσπιση μηχανισμού επίλυσης διαφορών. Επίσης για την Ευρωμεσογειακή Συμφωνία και για το μηχανισμό επίλυση διαφορών που εφαρμόζεται διαφορέ στο πλαίσιο εμπορικών διατάξεων ε, τη Ιορδανία και τέλο τη Αιγύπτου. Αυτέ είναι λοιπόν οι εμπορικέ συμφωνίε οι οποίε ε, όπου προβλέπονται δηλαδή διατάξει για την απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών και που βασίζονται ιδίω σε διπλωματικές προσεγγίσεις αυτές οι προσπάθειες επιλύσεως διαφορών όμως ε, μέχρι τώρα είναι αναποτελεσματικές διότι εύκολα μπορούν να μπλοκαριστούν από ένα ενδιαφερόμενο μέρος. Το Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσει με τους εταίρους της Ευρωμεσογειακής Ζώνης για να θεσπιστούν μηχανισμοί βασισμένοι στο μοντέλο της επίλυσης διαφορών των πιο πρόσφατων συμφωνιών και του μνημονίου που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Εν προκειμένου πρόκειται για τις χώρες Μαρόκο, Ιορδανία και Αίγυπτο. Εδώ απαιτείται τώρα η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν να μπορέσουν να ισχύσουν. Αυτές οι τρεις λοιπόν συμφωνίες είναι πολύ παρόμοιες και γι' αυτό θα τις συζητήσουμε όλες μαζί. Ο κάθε ένα εκ των εισηγητών βέβαια θα έχει, τον, θα έχει δυνατότητα να λάβει τον λόγο για την έκθεσή του. Έχουμε λοιπόν τρεις εισηγητές. Για το Μαρόκο είναι ο κύριος Κούτας, για την Ιορδανία ο κύριος Μενέντες και για την Αιγύπτο ο κύριος Σούστα. Όλοι είναι από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επιτρέψτε μου λοιπόν να δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Κούτας. Έχετε το λόγο, George. Ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε, Πρόεδρε. Η σύμφωνη γνώμη που ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρεται στην, στις διαπραγματεύσεις για την θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών με το βασίλειο του Μαρόκου. Η ε, πρόταση συμφωνίας έχει σκοπό να αυξήσει την ασφάλεια και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων με τη θέσπιση ενός μηχανισμού επίλυσης διαφορών με αποτελεσματικές διαδικασίες και με χρονικά όρια. Όπως είπατε πριν, για την ώρα η επίλυση διαφορών γίνεται μέσω διπλωματικών ε, ε, διάβλων και εύκολα μπορούν να βλοκαριστούν από κάποιο ενδιαφερόμενο μέρος. Εν προκειμένου, για την, στην προσπάθεια μάλλον αναβάθμισης των εμπορικών σχέσεων μέσα στην ευρωμισαγιακή ζώνη, θεωρήθηκε σωστό να υπάρξει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Στις 24 Φεβρουαρίου 2006 η Κομισιόν άρχισε διαπραγματεύσεις με τις ε, χώρες της Ευρωμεσογειακής Ζώνης για το θέμα αυτό. Οι διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο οδήγησαν εν τέλει σε σχέδιο συμφωνίας Αρχικά υποβλήθηκε αυτό στη ε, διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου το Δεκέμβριο 2009 στις Βρυξέλλες, βασισμένο στο ε, μοντέλο του ε, ΠΟΕ, ε, του μνημονίου του ΠΟΕ και βέβαια έχει προσαρμοστεί στο διμερές αυτό πλαίσιο. μετά από παραβίαση του δευτέρου τίτλου της συμφωνίας σχετικά με ε, προϊόντα αγροτικά και αλίας και με εξαίρεση των άρθρων anti-dumping. Προβλέπει την δυνατότητα να επιλύονται διαφορές μέσω διαιτησίας και διαμεσολάβησης. Υπάρχουν κανόνες για την διαφάνεια και συμμόρφωσης με το μνημόνιο, όπως είπα, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μενέντες για την Ιορδανία. Gracias, presidente. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, αυτά τα τρία, αυτές οι τρεις συμφωνίες συνδέονται μεταξύ τους και ο τρόπος με τον οποίο τα εξήγησε ο συνάδελφος κύριος Κούτας είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό. Άρα λοιπόν δεν έχω κάτι να προσθέσω γιατί το πλαίσιο αναφοράς είναι προφανέστατα το ίδιο. Θα ήταν λοιπόν τελείω ε, αδιανόητο να επαναλάβω εδώ τα όσα είπε ο συνάδελφος. Προσυπογράφω, λοιπόν τα δικά του σχόλια και φαντάζομαι ε, πως αυτά θα ισχύσουν και στην περίπτωση τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Όπω όπως ε, και στο άλλο θέμα το οποίο, με το οποίο ασχολήθηκα, που είναι οι κανόνες ε, για χώρα καταγωγής. Οι συνθήκες αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί έχουν σκοπό να τελειοποιήσουν την αρχική διαδικασία της Βαρκελόνης, η οποία οδήγησε στην Ένωση για τη Μεσόγειο σήμερα, γιατί για διάφορους λόγους υπάρχουν μία σειρά από ε, επιπλοκές ε, που μπορούν να ξεπεραστούν μόνο εάν εγκρίνουμε κοινά εργαλεία, κοινά μέσα. Διαφορετικά οι διαπραγματεύσεις καθυστερούν. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές, αλλά πρέπει να σας πω πως τα όσα έχουμε θεσπίσει είναι σε απόλυτη συμφωνία με τα όσα έχουμε ε, στον ΠΟΕ. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει καν μια υποψία σκιάς που να σκιάζει αυτή τη συμφωνία. Άρα δεν έχω κάτι παραπάνω να προσθέσω on Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αφού άκουσα το φίλο Εμίλιο, εγώ δεν έχω να προσθέσω πολλά, αλλά απλώς να θυμίσω ότι οι διαπραγματεύσεις με την Αίγυπτο για το μηχανισμό αυτό έχουν ε, ολοκληρωθεί το 2007. Είναι μια συμφωνία που ακολουθεί τα μοντέλα που ε, έχει συναυθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες χώρες αλλά και με την Διεθνή Οργάνωση για το Εμπόριο, ε, τον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου και γι' αυτό θα πρέπει να οριστεί το συλλογικό όργανο, η διαδικασία, μια λογική χρονική περίοδος για την εκτελήση των διορθωτικών μέτρων, των προσωρινών. Είναι δηλαδή ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι απαραίτητο στην πράξη όλα αυτά τα μέτρα να χρησιμοποιηθούν. Ε, όπως σε άλλες περιπτώσεις όπως με την Τουρκία δεν συνέβη πάντοτε. Η ευχή μας είναι λοιπόν να ξεπεραστεί η διπλωματική καθαρά ε, λύση και να βρεθούν πιο αποτελεσματικά μέτρα για να λύνονται ε, οι, τα προβλήματα και οι διαφορές. Τα υπόλοιπα συμφωνώ με τους προηγούμενους συνάδελφους. Ευχαριστούμε, ακούσουμε την Επιτροπή. Σοφία Μουνιός. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω. Νομίζω ότι όλα υπόθηκαν πια από τους προηγούμενους ομιλητές, από εσά και από τους τρεις εισηγητές. Και όπως είπατε, η δημιουργία αυτή των μηχανισμών επίλυσης διαφορών μέσα στις ε, συμφωνίες ε, σύνδεση και εταιρική σχέσει. Είναι πολύ σημαντικό βήμα στι μεσογειακέ μα σχέσει γιατί δείχνει ότι αναβαθμίζουμε τι συμφωνίε μα με αυτέ τι χώρε. Και αυτό που λέμε στις χώρε αυτές είναι ότι όταν δουλεύουμε παράλληλα προς ε, ένα βελτιωμένο προηγμένο στάδιο μαζί τους Οι καλοί κανόνε χρειάζονται και καλή διαδικασία ε, εφαρμογή επιβολής. Και αυτό κάναμε τώρα με τις χώρες αυτές. Αυτά έχω να προσθέσω στα όσα ήδη είπατε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε με τους ε, σκιώδες. Άλβες. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο και θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι οι συγητέ. Επιμένω λοιπόν πως το ΕΛΚ με ενθουσιασμό υποδέχεται την πρόταση αυτή της Κομισιόν για το μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Σας ευχαριστώ πολύ. Any other speaker? So there's a happy unanimity consideration of draft reports will take place next. Ευχαριστώ πολύ. Η κατάθεση των ε, η ψηφοφορία θα γίνει στις 26 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 21, Περιφερειακή Σύμβαση για τις Πανευρωμεσογειακούς Προτιμησιακούς Κανόνες Καταγωγής. Συγητής είναι ο κύριος Μενέντες από τους Σοσιαλιστές ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι το Δεκέμβριο πέρυσι η Υπουργοί Εμπορίου της Euromed ενέκριναν ένα σχέδιο σύμβασης για τους ευρω... ευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες για τους οποίους ζητά τη συνένεση του Κοινοβουλίου ή Κομισιόν. Η ιδέα της σύμβασης είναι να αντικαταστήσει την ε, διαδικασία που βασίζεται σε διμερή πρωτόκαλα από ένα μόνο νομικό μέσο υπό τη μορφή μιας περιφερειακής σύμβασης. Αρχικά η πρόταση και... Ε, ε, προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του έτους, αλλά οι συζητήσεις συνεχίζονται ακόμα στο Συμβούλιο και γι' αυτό το λόγο πιθανότατα δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί σε αυτό το διάστημα. Ενώ ε, περιμένουμε επισήμως να έρθει σε επαφή μαζί μας το Συμβούλιο, εμείς θα το συζητήσουμε και βεβαίως θα ε, μπει επισήμω στο πρόγραμμά μας από τη στιγμή που θα έχουμε την επίσημη απόφαση του Συμβουλίου. Μετά από αυτό το πρόλογο δίνω το λόγο στον Εμίλιο Μενέντε. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπα προηγουμένως, αυτή η πρόταση του Συμβουλίου που μας απασχολεί τώρα προσπαθεί με τον τρόπο της να διευκολύνει ε, την ε, δρομολόγηση των διαφορών διαδικασιών για την ε, λειτουργία της ε, Ένωσης της Μεσογείου, της Μεσογειακής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν τους κανόνες καταγωγής που είναι ένα εμπόδιο που πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεραστεί για να δημιουργήσουμε αυτή την ελεύθερη ζώνη εμπορίου μεταξύ Μεσογείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήμερα το πανευρωπαϊκό σύστημα για τη σώρευση των κανόνων καταγωγής έχει κατακλειστεί από με ένα τεράστιο αριθμό συμφωνιών, πρωτοκόλων κτλ. που ουσιαστικά δημιουργεί μια πολυσπερμία ε, ρητρών και διατάξεων, γιατί βέβαια εφόσον ένα κράτος υπογράψει με κάποια άλλο μια συμφωνία, μετά αυτό πρέπει να τοποθετηθεί και στις συμφωνίες της διμερής που έχει με τα υπόλοιπα κράτη, κάτι το οποίο δημιουργεί χάος. Άρα λοιπόν το Συμβούλιο προσπαθεί κάπως να συγκεράσει όλα αυτά τα στοιχεία, δηλαδή δημιουργήσει ένα μοναδικό νομικό μέσο, το οποίο επαναλαμβάνω θα μας ε, χρησιμεύσει για να κάνουμε κάποια πρόοδο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι πως βρισκόμαστε εν αναμονή της ε, επίσημης πρότασης του Συμβουλίου, γιατί το θέμα που συζητάμε έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί στην 9 Δεκεμβρίου από τους Υπουργού Εμπορίου στις Βρυξέλλες, όμως ακόμα δεν έχουμε την γνωμοδότηση του Συμβουλίου. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε το θέμα σε ένα πρώτο στάδιο, παρόλο που δεν έχουμε επίσημη θέση του Συμβουλίου, γιατί πιστεύω πως δεν θα πρέπει τουλάχιστον να μας δημιουργήσει κάποια εμάς προβλήματα, σε καμία από τις πολιτικές ομάδες, τουλάχιστον όχι ουσιαστικά προβλήματα. Και επειδή εμείς θα συμφωνήσουμε γρήγορα το θέμα αυτό, θα μπορέσει και το εμπόριο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ. Να ακούσουμε λοιπόν την Επιτροπή. Ποιο θα λάβει το λόγο εκ μέρου τη. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει κάθε προσπάθεια ώστε η συμφωνία αυτή να λάβει σάρκα και ωστά. Η αρχική μας πρόθεση ήταν να είναι σε ισχύ από την αρχή του επόμενου έτους, όμως ε, λόγω των ε, προβλημάτων με τον ορισμό του κοσυφοπεδίου θα έχουμε κάποια καθυστέρηση. Ο λόγος για τον οποίο η σύμβαση αυτή είναι σημαντική για τις ευρωμεσογειακές εμπορικές σχέσεις είναι πως για τους εταίρους μας στη νότια πλευρά της Μεσογείου είναι πολύ σημαντική, αλλά και γιατί τα Δυτικά Βαλκάνια εδώ και τέσσερα χρόνια περιμένουν να συμπεριληφθούν στο ε, πανευρωπαϊκό σύστημα των κανόνων καταγωγής. Έχουμε λοιπόν μια προβληματική κατάσταση η οποία θα μας ξαναπασχολήσει στα, στη διάρκεια, στο διάστημα που θα διανύσουμε μέχρι τις 11 Νοεμβρίου που θα γίνει η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη Υπουργών Εμπορίου και πάλι θα έρθουν οι Υπουργοί Εμπορίου της Νοτιού Μεσογείου και θα μας ρωτήσουν πώς προχωράτε με τη συμφωνία αυτή. με τη συνθήκη αυτή. Ο εισηγητής έκανε μια πολύ σωστή παρουσίαση. Είναι σημαντική γιατί θα ε, ε, διευκολύνουμε την αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής και γιατί τα μέσα που έχουμε μέχρι σήμερα και οι συνθήκες που έχουμε είναι κάπως απαρχαιωμένες και λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης που έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε την έγκρισή της και να ε, διευκολύνουμε όλες αυτές τις ε, διαδικασίες. Αυτό είναι ένα αίτημα ηχηρό από τους γείτονές μας ε, στο Νότο και βέβαια έχουμε και το θέμα, όπως σας είπα, των Δυτικών Βαλκανίων. Ελπίζω πως σύντομα θα είμαστε σε θέση να ξεμπλοκάρουμε τις συζητήσεις για το πολιτικό ζήτημα που ε, μπλοκάρει την έναρξη των, αυτής της ε, συνθήκης και πώς θα την έχουμε στα χέρια μας το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Υπάρχουν ε, συμβολές. Χέλμουτ Σόλτς. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τώρα για τις ιδιαίτερες σχέσεις της Ένωσης με το Μαγκρέμπ σχετικά με τον προτινόμενο κανονισμό θα προβλέπει ο κανονισμός μια μεικτή επιτροπή με το δικαίωμα να αποδέχεται νέα μέλη στο καθεστώς αυτό. Και αυτές ε, θα επιτρέπονται αποκλειστικά για τον χώρο της Μεσογείου. Δεύτερο, αυτή η μεικτή επιτροπή θα δρά ε, σε συνθήκες ομοφωνίας. Το άρθρο 5 4 λέει ότι δεν επιτρέπεται ένα μέλος να μπλοκάρει την είσοδο νέου μέλους. Ερώτηση προς την Κομισιόν. Ποια είναι η αιτιολόγηση αυτής της εξαίρεσης. Τρίτη ερώτηση. Προβλέπει ο κανονισμός να ε, ε υπάρχουν τον στον κανονισμό για προϊόντα που έρχονται από την Παλαιστίνη και να ε, φέρουν την ονομασία αυτή προέλευσης. Κάτι που θα αποτελούσε μια σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει την αγορά της δηλαδή σε προϊόντα made in Palestine, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον Παλαιστινιακό λαό την ευκαιρία να μπορέσουν να ζήσουν από την δική τους παραγωγή. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει, υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε κάτι να απαντήσετε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Δυστυχώς οι συνάδελφοί μου που είναι οι εμπειρογνώμονες της ΙΤΑΞΟΥΝΤ δεν έχουν φτάσει ακόμη. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Ναι, εδώ βλέπω πράγματι ότι η Κομισιόν πρόκειται να εκπροσωπηθεί από άλλους. Καταλαβαίνω λοιπόν ποιο πρόβλημα έχετε. Αλλά παρόλα αυτά αν μπορείτε, καλά, η ε, εκπρόσωπη της Κομισιόν θα προσπαθήσω. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση νέων μελών και το γεγονός ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο μπλοκαρίσματος, νομίζω ότι η διατύπωση που περιλαμβάνεται στην συμφωνία ήταν αντικείμενο προσεκτικής διαπραγματεύσεως για να αποφευθεί πράγματι τέτοιο ενδεχόμενο αποκλεισμού. Η ιδέα ήταν δηλαδή να υπάρξει μια συνένεση μείον ενός, μείον μιας χώρας. Τέθηκε μια ερώτηση ακόμη. σχετικά με τους παράνομους επικισμούς στην Παλαιστίνη η συμφωνία δεν αλλάζει την ισχύουσα κατάσταση. Τα προϊόντα αυτά ε, ε, εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ισχύ τεχνικών ε, ρυθμίσεων που σημαίνει ότι δεν εποφελούνται από τις προτιμήσεις, δεν απολαμβάνουν δηλαδή προτιμήσεις. Καμιά φορά εδώ υπάρχει σύγχυση με τους κανόνες επισήμανσης, labeling rules. Η συμφωνία αυτή δεν πρόκειται να τροποποιήσει την κατάσταση αυτή. Δεν πρόκειται να διασαφίζει ποια προϊόντα παράγονται στους επικισμούς και ποια στο Παλαιστινιακό έδαφος. Η ε, Παλαιστινική Αρχή δεν έχει ακόμα εφαρμόσει το Ευρωμεσογειακό Πρωτόκολλο. Θα το πράξει αυτό όταν θα ε, συμμετάσχει στην συμφωνία και θα έχει την δυνατότητα να συμμετάσχει στο εμπόριο με άλλε χώρε τη Νότια Μεσογείου, με την οποία έχει συμφωνίε. και επομένω τώρα ε, η Ορδανία, Τουρκία και Ισραήλ, στο μέλλον αυτό θα περιλαμβάνει και το Αγαδίρ, γιατί οι χώρες αυτές είναι υποψήφιες για να συμμετάσχουν στη Συμφωνία Αγαδίρ και αυτό θα συμβεί μάλλον σύντομα. Άρα, η Συμφωνία δεν πρόκειται να προσφέρει νέα στοιχεία σε ό,τι αφορά την επισήμανση των ε, συγκεκριμένων προϊόντων, θα επιτρέψει όμως καθαρά παλαιστινιακά προϊόντα ε, να εποφελούνται από την συσσόρευση ε, και άλλων ευκαιριών που δίνονται από άλλα πάνελ της ευρωμεσογειακής ζώνης. Μενέντες θέλετε να μιλήσετε. Όχι, όχι, είναι σαφή τα πράγματα. Θα περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Σημαντικό πράγματι. Και ας προχωρήσουμε τώρα στο 22. Ε, Point was moved to the afternoon. Το σημείο 22 έχει μεταφερθεί για την απογευματινή συνεδρίαση, οπότε πάμε στο 23 γιατί έγινε εκεί μια ανταλλαγή. Φορολογία και ανάπτυξη, συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα. Έχουμε γνωμοδότηση εδώ. της Επιτροπής Ανάπτυξης που είναι αρμόδια επί της ουσίας και συντάκτης ε, γνωμοδότησης είναι η Μαριέλ Τεσσαρνές. Και εδώ θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης της γνωμοδότησης μάλλον. Είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της ΔΕΒΕ για τη φορολογία και την ανάπτυξη μετά από μια ανακοίνωση της ε, Κομισιόν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Εμείς ε, στις 9 Δεκεμβρίου θα ε, ψηφίσουμε και η ανακοίνωση της Κομισιόν προτείνει τρόπους με, τον οποίο, με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες ώστε να θεσπίσουν αποτελεσματικά και δίκαια φορολογικά συστήματα ώστε να κινητοποιηθούν οι χώροι οι πόροι μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. Εμείς αποφασίσαμε να συμβάλλουμε με μια γνωμοδότηση και δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας Μαριέλ Ντεσαρνέζ από την ομάδα ALDE. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πιστεύω πως αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών με τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει επιπτώσεις ορισμένες φορές θετικές, ορισμένες αρνητικές. Ιδιαίτερα όσον αφορά την μείωση των δημόσιων εσόδων. Όντω η κατάργηση των τελωνιακών δασμών αποτελεί μια μεγάλη απώλεια εσόδων και άρα μια πιθανή μείωση των κοινωνικών δαπανών ή των δυνατοτήτων επενδύσεων, των επενδυτικών μάλλον δυνατοτήτων των χωρών αυτών. Επίση, θα πρέπει να προσθέσουμε και δεν το λέμε συχνά ότι η κατάργηση των ανταλληνικών δασμών έχει επίση επιπτώσει και αντίκτυπο στου άλλου φόρου. Γιατί οι φόροι στα εισαγόμενα προϊόντα όπω το ΦΠΑ ε, υπολογίζονται μέσα στην αξία, ε, πάνω στην αξία μάλλον του αγαθού μετά από την εφαρμογή του τελωνιακού δεσμού. και γι' αυτό και η, φορολογική διαχείριση είναι για μα ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Νομίζω πω είναι ζωτική σημασία καλύτερα να χειριστούμε την κατάργηση των φορολογικών δασμών, ίσω να γίνουν των τελωνιακών δασμών, συγγνώμη, ίσως να γίνει αυτό σταδιακά και παράλληλα να γίνει μια φορολογική μεταρρύθμιση που θα επιτρέψει να κινητοποιηθούν αντισταθμιστικά έσοδα. Για να φτάσουμε σε αυτό το στόχο πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε στήριξη για την φορολογία αυτών των χωρών, για την απαραίτητο, αλλά και να διευκολύνουμε τις εφορίες ώστε να έχουν μια καλή φορολόγηση. Πολύ συχνά η φορολογική νομοθεσία είναι εξαιρετικά περίπλοκη, οπότε θα από τη μια πλευρά την φοροδιαφυγή αλλά και την διαφθορά. Γιατί κάποιες φορές ε, γίνεται η συλλογή των φόρων με ε, διακρίσεις όπως ε, για να το πω έτσι πράγμα το οποίο θα ρίνει την ε, διαφθορά. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρες αυτές να βρουν μια νέα, ένα νέο έσοδο για να αντισταθμίσουν τις απώλειες που έχουν, τις ζημιές που έχουν. Καταρχήν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διευρυνθεί η φορολογική βάση με ένα αρχικό φόρο χαμηλό και έπειτα να, αποκλειστούν κάθε, να αποκλειστεί κάθε είδος εξαιρετικού και φορολογίας για τις εξορρυκτικές βιομηχανίες. Εκεί υπάρχει πολλά που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά μέσα στο πλαίσιο της καλής διαχείρισης και διακυβέρνησης, αλλά να αποφύγουν, να αποφευχθεί και η διαρροή των κεφαλαίων προς τους φορολογικούς παραδείσους, που είναι καθήκον του Κοινοβουλίου ως διεθνούς οργανισμού. Και έπειτα, επίσης, τοπικά θα πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο φορολογικό σύστημα με μεγαλύτερη ε, νομική ασφάλεια που συχνά δεν υπάρχει. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικέ και βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή στην καινοτομία και στην μεταφορά γνώσεων ώστε πραγματικά να οθήσει την ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες. Ε, εξίσου πιστεύω πως είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύστημα ανεξάρτητο για τον έλεγχο που θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο το συγκεκριμένο της κατάργησης των ε, τελωνιακών δασμών όχι σε μεγάλα μπλοκ, σε μεγάλες περιοχές αλλά ανά χώρα πραγματικά και θα μετρήσει επίσης την αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων των φορολογικών και την αποτελεσματικότητα της φορολογικής αυτής της χώρας είναι πολύ πολύ σημαντικό. Σε αυτά περιορίζομαι σε αυτή τη γνωμοδότηση. Νομίζω πως είναι απαραίτητο να εισαχθεί μια ρήτρα που θα προβλέπει την υποχρεωτική εξέταση, αναθεώρηση κάθε τέτοια συμφωνία μετά από πέντε χρόνια και την ενδεχόμενη τροποποίησή της, λαμβάνοντας υπόψη την, ε, την αξιολόγηση που θα γίνει. Αυτές είναι χοντρικά οι γραμμές που θελήσαμε να κρατήσουμε μέσα στην γνωμοδότηση αυτή και φυσικά θα είμαι στη διάθεση των συναδέλφων να τους ακούσω είτε προφορικά είτε μέσω των τροπολογιών τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ε, δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν που είναι ο Μάρτιν Ζαουραλόβα. Όχι, δεν είμαι ο, Μαρτίν Ζαολάβα ή Μαρτίν, <laughs> όπως βλέπετε, που δεν μπόρεσε να φτάσει ακόμη. Οπότε θα απαντήσω στην θέση της. Σας παρακαλώ πείτε μας το όνομά σας. Ζόρζα Χαραβαλέ. Βασικά συμφωνούμε με τις ε, κύριες αρχές της νομοδότησης. Να σας πω μόνο ένα θέμα ε, που αφορά την ε, κατάργηση των δασμών. Ότι αυτό, λέτε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει με σταδιακό τρόπο και σε αυτό συμφωνούμε μαζί σας γιατί θα πρέπει να δούμε ότι ε, εκεί όπου γίνεται αυτό ε, γίνεται σε σχέση με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές της Ένωσης δεν είναι για όλα τα προϊόντα υπάρχουν ξερέσεις που φτάνουν μέχρι το 20% της κάλυψης ε, όσον αφορά τα προϊόντα στις συμφωνίες αυτές και έπειτα για τα υπο... τους υπόλοιπους δασμούς για τα υπάρχοντα προϊόντα δηλαδή για το 80% των δασμών που θα καταργηθούν υπάρχει μια σταδιακότητα που προβλέπεται μέχρι 20 και 25 χρόνια μπορεί να φτάσει και το έχουμε δει ήδη στις συμφωνίες που έχουμε διαπραγματευτεί μέχρι στιγμής. Ε, τώρα όσον αφορά την αρχή τη αξιολόγηση των συμφωνιών μετά από πέντε χρόνια, αυτή είναι μια αρχή που ήδη ισχύει. Ε, θυμάστε ότι έγινε αυτό για την ακτή του Αλεφαντοστού και μπορεί να έχετε βέβαια και άλλες παρατηρήσεις να κάνετε με την Γενική Διεύθυνση ΔΕΒΕ. Ε, αυτά είχα να πω εγώ για τις δικές μας αρμοδιότητες. Θα ζητήσω από την Κομισιόνα να μην αλλάζει έτσι προσδόκητα τους εκπροσώπους της αυτές τις συνεδριάσεις. Ας ε, συζητήσουμε λοιπόν το θέμα. Αρχίζουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ο Δανιέλ Κάσπαρη από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Είναι καλό που εγκύπτουμε στο θέμα εδώ ως Επιτροπή. Κατ' επανάληψη έχουμε σημειώσει ότι σε ό,τι αφορά την ίσπραξη φόρων πολλές χώρες του κόσμου έχουν προβλήματα, για παράδειγμα αφρικανικές χώρες. Εξαίρετα δεξίγει αυτά η εισηγήτρια στην εκθεσή της δείχνει σαφώς τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει ένα ε, ατελέσει και ανύπαρκτο ε, σύστημα φορολογικών εισπράξεων. Χαίρομαι που κάνει και προτάσεις η εισηγήτρια. Εμείς έχουμε λίγες συμπληρώσεις να κάνουμε, τις οποίες ελπίζω να εξετάσει ε, με θετικό πνεύμα η εισηγήτρια, να δούμε πώς θα καταφέρουμε η συζήτηση αυτή να περιστραφεί γύρω από ένα καλό και χρήσιμο φορολογικό σύστημα και η συζήτηση αυτή να προωθηθεί και σε άλλα θεσμικά όργανα. Δηλαδή, Μπορούμε να θέσουμε το θέμα αυτό περισσότερο και στις ημερήσεις διατάξεις της Ισομερούς Συνελεύσεως των χωρών ΑΚΕ. Επίσης στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Είναι σαφές ότι η κατάσταση στην Αφρική είναι πολύ δύσκολη. διότι αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν φόρους είναι και αυτοί που καλούνται να τροποποιήσουν το σύστημα. Δεν θα είναι λοιπόν ιδιαίτερα ενθουσιώδης υπέρ μιας αλλαγής αλλά βλέποντας σε ποιες δραματικές δυσχέρειες σε ποιες μάλλον δραματικές δυσχέρειες οδηγεί ε, το σύστημα, τα συστήματα ή τα ατελή ή ανύπαρκτα αυτά συστήματα προς το συμφέρον μιας βιώσιμης ανάπτυξης και μιας ε, ε, ευημερίας βασισμένης στην ανάπτυξη αυτή είναι απόλυτα απαραίτητο να συζητηθούν και να προωθηθούν. Σας ευχαριστώ. Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω πρώτα πρώτα την εισηγήτρια για την προσέγγιση που επέλεξε για το θέμα στην γνωμοδότησή της. Πρόκειται πράγματι για πρόβλημα μεγάλης βαρύτητας. Η κατάσταση που συνδέεται άλλωστε με την οικονομική κατάσταση των χωρών ΑΚΕ και είναι πολύ θετικό το ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. Εγώ επίσης θεωρώ τον συνδυασμό αυτού του φορολογικού dumping από τη μια μεριά και την ανάπτυξη σε άλλες χώρες από την άλλη μεριά, τα θεωρώ αυτά ως μια πρόκληση που πρέπει να μας απασχολήσει, να δούμε δηλαδή εάν στις θέσεις που λαμβάνουμε και ως Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, αν πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα και την ευθύνη των φορολογουμένων. Άρα και οι επενδυτές πρέπει να καταστήσουν σαφές και διαφανές ότι πληρώνουν φόρους και ότι είναι υπέρ ενός υπεύθυνου φορολογικού συστήματος στις χώρες αυτές. Δεύτερο, να εγκαταλείψουμε την πρακτική που βλέπει επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων από τις ευρωπαϊκές χώρες να συμβάλλουν στην διαφθορά στις αφρικανικές χώρες κάνοντας ε, για να μην πω δωροδοκίες αλλά πολύ γενναιόδορες προσφορές ας το πω έτσι λοιπόν αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πάυσει αυτή η δραστηριότητα. Τέλος επίσης το γεγονός ότι χρήματα των φορολογουμένων των ίδιων των αφρικανικών χωρών καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους και αυτός ο συσχετισμός λοιπόν πρέπει να τεθεί επιτάπητος. Τέταρτο, εμείς οι ίδιοι πρέπει να εγκύψουμε ξανά στο θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης, του δίκαιου χαρακτήρα δηλαδή των φορολογικών συστημάτων, ώστε να αποφεύγεται το φορολογικό dumping. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε άλλους λοιπόν ομιλητές που μας θέλουν να πάρουν το λόγο. Θα δώσω το λόγο στην κυρία της Αρνής για να σχολιάσει τα όσα άκουσε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους που έλαβαν το λόγο και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν. Νομίζω πως η ορθή χρηστή οικονομική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντική και η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος στην Αφρική είναι σημεία τα οποία πρέπει να προωθήσουμε ε, και κυρίως υπέρ των απόρων και των αδυνάμων. Με τα όσα είπε λοιπόν ο κύριος Κασπάρη συμφωνώ, με τα όσα είπε ο κύριος Σόλς συμφωνώ, η ορθή φορολογική, χρηστή φορολογική διαχείριση θα πρέπει να ισχύσει όχι μόνο για τα αφρικανικά κράτη, αλλά και για τα ευρωπαϊκά. Θα πρέπει λοιπόν αυτές τις αρχές να τις εφαρμόσουμε και οι ίδιοι πριν ζητήσουμε να τις εφαρμόσουν οι υπόλοιποι. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό αυτό και συμφωνώ και με τα όσα είπατε για τους φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει να το επενθυμίσουμε σε αυτή τη γνωμοδότηση και νομίζω πως θα πρέπει να το επενθυμίσουμε και σε άλλες συζητήσει που κάνουμε και κυρίως στην ε, G20 ε, γιατί εκεί έχουν συζητηθεί πολλά ε, ήδη εδώ και δύο χρόνια για τους φορολογικούς παραδείσους και ακόμα δεν έχουμε κάνει τίποτα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα αυτό. Τώρα, για την σταδιακή εφαρμογή, μιλήσατε και εσείς για το θέμα αυτό, για την κλιμάκωση, νομίζω είναι σημαντικό να δούμε την αρχή της αξιολόγησης, έτσι ώστε να γίνει μια καλή αξιολόγηση χώρα-χώρα για να λάβουμε υπόψη τα θέματα αυτά, αλλά με πιο πολιτικό τρόπο, όχι τόσο διοικητικό. Euh, e για να δούμε λοιπόν αν μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές και αν δεν το κάνουμε ε, νομίζω ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Αφού θέλουν να υπογράψουν μαζί μας, ας φανούμε τουλάχιστον ευφυείς στις προσπάθειες που θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ. Να σας πω λοιπόν πως η έγκριση της, ε, του σχεδίου γνωμοδότησης είναι για το Δεκέμβριο, άρα λοιπόν έχουμε μέχρι τις 28 του μηνός για να υποβάλουμε τροπολογίες στις 6 ώρα το απόγευμα του τρέχοντος μηνός. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της ε, σημερινής μας πρωινής συνεδρίασης και ο λόγος για τον οποίο τελειώνουμε τόσο νωρί είναι πως έχουμε αναβάλει τρία θέματα. Μία πολύ σημαντική συζήτηση για την στρατηγική για το 2020 στην οποία είχαμε διαθέσει μία ώρα, όπως επίσης και την δημόσια κρόση για τις επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω πως στο μέλλον θα είμαι λιγότερο, λιγότερο γενναιόδωρος όταν μου ζητάτε κάποια αναβολή. Να κάνω και δύο ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα πως το απόγευμα θα συνειδριάσουμε σε άλλη αίθουσα, όχι εδώ, στην 5G2 και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράψει πως η σειρά των συζητήσεων το απόγευμα είναι η εξής. Σημείο 22. Σημείο 22. Δασμολογική ατέλεια για συγκεκριμένα φαρμακευτικά δραστικά συστατικά. Μετά το 24, αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία των αγορών. Το 26, απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Το 27, κανονισμός που θεσπίζει τους κανόνες και τις γενικές αρχές για την Επιτροπή και τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. 28, μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης. 29, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Και το 30, ανταλλαγή απόψεων όσο αφορά όσον αφορά τι εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ινδίας εν ώψη της διάσκεψη κορυφη Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ινδίας. Πολύ σημαντικά θέματα το απόγευμα. Αλλά έχουμε αλλάξει, όπω είδατε, λίγο τη σειρά. Θα τα δούμε μετά το μεσημεριανό γεύμα. Σα ευχαριστώ πολύ.